Proszę ε, Państwa, jeszcze chwilę zajmiemy się budżetem. Μισό λεπτό ακόμα, συνάδελφοι, για τον προπολογισμό πάντα. Πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση Σουριάν και Μάνκα για το σχέδιο Γενικού Προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2010, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο, σε όλα τα τμήματά του. Ψηφίζουμε την τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τέταρτη παράγραφος θα ψηφιστεί σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η παράγραφος, το πρώτο τμήμα της τέσσερα. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα της παράγραφου τέσσερα. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ε, ψήφισαν υπέρ 320, κατά 236, 10 αποχές. Εγκρίνεται. Χρειαζόμαστε τώρα απλή πλειοψηφία, γι' αυτό εγκρίθηκε. Τροπολογία 1. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 314 υπέρ, 237 κατά, 20 εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ο κύριο Σούριαν υποβάλλει μια προφορική τροπολογία και του δίνω το λόγο. Κύριε Σούριαν, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, προτείνεται οι τροπολογίες 3 ή 7 που είναι ίδιες να ψηφιστούν κατά τρία τμήματα. Η προφορική τροπολογία αλλάζει το δεύτερο τμήμα. Γιατί το αρχικό κείμενο ανέφερε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής. Εν τω μεταξύ ωστόσο το Συμβούλιο αποφάσισε επί του θέματος αυτού. Διαβάζω λοιπόν τη νέα πρόταση. Πιο συγκεκριμένα. Σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να συμβάλλουν σε αυτό το, ε, το, τη χρηματοδότηση ταχεία μορφή με 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίω από τα έτη 2010 στο 2012. Υπογραμμίζει ωστόσο την ανάγκη ενημέρωση για τη συμμετοχή και τη συνεισφορά του προπολογισμού τη Ένωση κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012. Αυτή είναι η προφορική τροπολογία. Η πρότασή μου είναι να υπερψηφιστούν και τα τρία τμήματα. Να ψηφίσουμε υπέρ και για τα τρία τμήματα. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος ο οποίος ε, είναι αντίθετος με την προφορική αυτή τροπολογία. Δεν βλέπω αντιρρήσεις, άρα μπορούμε να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε κατά τρία τμήματα όπως σας είπα. Με ονομαστική ψηφοφορία κάθε τμήμα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 525 υπέρ, 25 κατά. 11 αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. με την προφορική η τροπολογία. Αρχίζουμε να ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 515 υπέρ, 28 κατά, 17 αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Εγκρίνεται η ψηφοφορία. Α, άρχεται η ψηφοφορία, συγγνώμη. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 515 υπέρ, 29 κατά, 18 αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εψήφισαν υπέρ 483, κατά 48, αποχές 32. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια ξανά προς τους εισηγητές, προς όλους μας, τις επιτροπές που ασχολήθηκαν με τον προϋπολογισμό. Ολοκληρώθηκε έτσι η ψηφοφορία του προϋπολογισμού. Κύριε Σούριαν, κύριε Μάνκα, συγχαρητήρια, μπράβο, πολύ καλά και με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και καλές διακοπές για τις τρεις αυτές εβδομάδες. Ξέρετε ότι κατά το προσεχές έτος μας περιμένει πολλή δουλειά και στις 12 Ιανουαρίου θα σας προσκαλέσω σε ένα κοκτέιλ για να γιορτάσουμε το νέο έτος και την ε, συνθήκη της Λισαβόνας που τέθηκε σε ισχύ. Ευτυχές στο νέο νέο έτος. Γεια σας. Okay, the next item is... Επόμενο σημείο είναι ψηφοφορία επί πέντε προτάσεων ψηφίσματος ε, για το νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση στα έγγραφα μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκη της Λισαβόνα. Κύριε Μπουζούτιλ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην ε, λίστα ψηφοφορία του ΕΛΚΑ έχει γίνει ένα λάθο. Να επισημάνω για του συναδέλφου λοιπόν ότι στι δύο ξεχωριστέ ψηφοφορίε το πρόσημο είναι συν. Επαναλαμβάνω για τις δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες που υπάρχουν, το πρόσημο είναι θετικό, συν. Δεν ξέρουμε, δεν ακούσαμε από την αρχή, το ήταν εκτός μικροφώνου το σχόλιο, είπε γιατί πρέπει να ακούμε αυτά που πρέπει να ψηφίσει το ΕΛΚ. Ήταν ε, το σχόλιο. Λοιπόν, η πρόεδρος ε, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται το 1 Χωριστή ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται και αυτό. Συνολικά η πρόταση ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα πέντε προτάσεις ψηφίσματος ε, για την περάσπιση αρχής επικουρικότητας. Κύριε Σούλτς. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Να επαναλάβω Χαίρομαι κυρία Πρόεδρε που τόσο έντονα ξυπνάω κάθε φορά του συναδέλφου και δεν του αφήνω να βαριέται και βοηθάει και την κυκλοφορία του αίματο. Ζητάω λοιπόν άλλη μια φορά βάση του άρθρου 177 παραγράφου 4 να αναβληθεί ε, η ψηφοφορία και να ελεγχθεί η παραδεκτότητα του ψηφίσματος. Έκανε την πρόταση το κύριο Σούλτ. Θα ακούσουμε έναν ομιλητή υπέρ και έναν ομιλητή κατά τη πρόταση του κύριου Σούλτ. Ποιο θέλει να μιλήσει υπέρ. Κατά. Ποιο θέλει να μιλήσει. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε. Το διαδικαστικό επιχείρημα που τέθηκε θα ήθελα να πω το εξή. Έχουμε και την έκθεση Κάσμαν, όπου εμεί ω ε, ε, κοινοβούλιο κάνουμε μία έκθεση για μία τρέχουσα νομοθετική διαδικασία και μα είπαν ότι δεν επιτρέπεται. Αυτό παρόλα αυτά οι σοσιαλιστέ επέμειναν όμω να προχωρήσουμε. Να πω ότι όταν, μιλάμε, όταν μιλήσαμε για την ελευθερία τη έκφραση στην Ιταλία, μα είπε ο Επίτροπο ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα. Και παρ' όλα αυτά οι σοσιαλιστέ επέμεναν να συνεχίσει η συζήτηση. Ε, λοιπόν, κυρίε και κύριοι, Όποτε ταιριάζει δηλαδή στους σοσιαλιστές δεν έχουμε αρμοδιότητα και όποτε δεν τους ταιριάζει έχουμε. Ε, δεν θα έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτό το επιχείρημα. Το δεύτερο επιχείρημα ωστόσο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σχετικής σύμβασης είμαστε αρμόδιοι. Θα ήθελα να σημειώσω ότι με τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας η Ένωση θα προσχωρήσει στη σύμβαση αυτή. θα πρέπει να το συζητήσει το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Γιαφόσον μπορεί να το συζητήσει το Ιταλικό Κοινοβούλιο, μπορεί να το συζητήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρίτο επιχείρημα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Τελευταίο επιχείρημα, Πρόεδρε. Τελευταίο. Κυρία Πρόεδρε, δεν είμαστε νομικοί, είμαστε πολιτικοί. Και αυτό το, αυτή η δικαστική απόφαση επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το ψηφίσουμε σήμερα. Θα ψηφίσουμε λοιπόν επί της πρότασης αναβολής. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Καλύτερα να το ελέγξουμε, θα ήταν πιο ασφαλές αυτό. Άρχεται λοιπόν ο ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψήφισαν όλοι. The vote is now closed. Πέρασε της ψηφοφορίας. Έγινε δεκτή η πρόταση. Επόμενο λοιπόν θέμα είναι η κατάσταση στη Λευκορωσία Νομίζω στην παράγραφο 17 έχουμε προφορική τροπολογία. Yes, thank you, Madam Chair. The sense of this... Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση για πρόσφατες ε, περιπτώσεις καταστολής στη Λευκορωσία. Ο στόχος μου είναι απλά να προσθέσουμε το όνομα ενός νέου ακτιβιστή, ο οποίος απήχθη στις 6 Δεκεμβρίου. Να προσθεθεί λοιπόν το όνομά του στον κατάλογο των ονομάτων που έχουμε σε αυτό το σημείο. Άρα μετά την αναφορά Σμίτσερ Δασκεβίτς να προσθέσουμε και Γιάουφε Νάχελ στις 6 Δεκεμβρίου 2009. Δηλαδή να προσθέσουμε ένα ακόμη άτομο στον κατάλογο που υφίστανται αυτές τις παρενοχλήσεις από την ε, λευκορωσική κυβέρνηση. Υπάρχουν αντιρρήσεις, λέει πρόεδρος, προς την προφορική τροπολογία αυτή. Από ό,τι φαίνεται όχι. Θα ψηφίσουμε λοιπόν την τροποποιημένη παράγραφο. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την κοινή πρόταση ψηφίσματος. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενο σημείο είναι έξι προτάσεις ψηφίσματος ε, για τη βία στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό στο κοινό ψήφισμα. Έχουμε πέντε πολιτικέ ομάδε. Τροπολογία 1, ψήφι υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Τροπολογία 2, ψήφι υπέρ, κατά, απόχέ. επίσης απορρίπτεται. Τροπολογία 3, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Με ονομαστική ψηφοφορία τώρα θα ψηφίσουμε την παράγραφο 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται παράγραφος 9. Τροπολογία 4 τώρα, επίσης με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται τροπολογία 4 και τώρα θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο του κοινού ψηφίσματος. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και έτσι ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες. Ευχαριστώ.